στρατηγική συνεργασία για την καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και της Ευρωπόλ. Θα δώσω το λόγο. Τέσσερα λεπτά στους δύο συγκητές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το κείμενο το οποίο συζητούμε αναφέρεται σε μια συμφωνία μεταξύ της Europol και των Ηνωμένων Αραβικών Εμβυράτων για την ε, στρατηγική συνεργασία στην καταπολέμηση του σοβαρού ε, οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Λόγω της ιδιαίτερης ε, στιγμής πρέπει να επικεντρώσουμε όλες τις προσπάθειές μας για να αντιμετωπίσουμε εγκληματικές ενέργειες που είναι ε, κατά των ε, προσωπικών ε, και οικονομικών συμφερόντων των πολιτών μας. Αυτό επίσης και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε οι δράστες να μπορούν να διώκονται από τη δικαιοσύνη. Σήμερα το Συμβούλιο ενέκρινε εν αναμονή της, προ... της πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την συμφωνία η οποία θα δημιουργήσει και θα ενισχύσει τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ε, για την ε, οργανωμένο έγκλημα μέσω της ανταλλαγής ε, πληροφοριών για συγκεκριμένες εξειδικευμένες γνώσεις. Πρόκειται για μια στρατηγική συμφωνία και όχι επιχειρησιακή και επομένω αποκλεί την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αρχίζουν να μετατρέπονται σε κόμβο οργανωμένου εγκλήματος, είναι χώρος προερισμού δραστών ε, και εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα απάτη ΦΠΑ, ε, νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων και είναι προφανές ότι ε, η ενίσχυση αυτής της συνεργασίας θα ενισχύσει και το ρόλο της Ευρωπόλ για την επίλυση ε, υποθέσεων που περιλαμβάνουν περισσότερο του ενός κρατών μελών, δύο και παραπάνω. Θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα μόνο μέσω διεθνούς συνεργασίας. Ε, με βάση λοιπόν τα όσα σας είπα και λαμβάνοντας υπόψη και τους όρους συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην διαδικασία που προβλέπεται σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, υπέβαλα μια έκθεση η οποία υποστηρίζει την απόφαση του Συμβουλίου να δώσει την έγκρισή, της, την έγκρισή του για τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπόλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα θα μπούμε στη διαδικασία Catch the Eye. Thanks. And now there are Υπάρχουν ε, τρεις ομιλητές. Ο κύριος Μαριάς πρώτος θα μιλήσει. Κύριε Πρόεδρε, περισσεύει η διγλωσία στο ζήτημα του χτυπήματος της τρομοκρατίας, ιδίως εν ώψη της στρατηγικής συνεργασίας των Ηνωμένων Αραβικών Ευρυμεράτων με την Europol. Και αυτό γιατί είναι γνωστό ότι εκτός από την Τουρκία υπάρχουν συγκεκριμένες αραβικές χώρες που ενισχύουν τον ΤΑΕΣ. Έτσι στις 16 Νοεμβρίου ο Βρετανικός guardian η γνωστή εφημερίδα παρουσίασε έγγραφο του state department των ηνωμένων πολιτειών που αποκαλύπτει τις οικονομικές σχέσεις των τζιχαντιστών με τη σαουδική αραβία άλλες αραβικές χώρες στις οποίες συμπεριλαμβάνει και τα ηνωμένα αραβικά εμιράτα. επομένως για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας του Ντάις πρέπει να κοπεί ο ομφάλιος λόρος μεταξύ της τρομοκρατίας και του χρήματος. αν τα αραβικά εμιράτα θέλουν να συμβάλλουν στο χτύπημα της τρομοκρατίας πρέπει να δεχτούν σε πρώτη φάση τους χιλιάδες πρόσφυγες από το ιράκ και τη συρία που έχουν κατακλείσει την ελλάδα και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. διαφορετικά όλα τα άλλα είναι μια φτηνή πολιτική κατανάλωση και προπαγάνδα προκειμένου να αποτελέσουν φύλλο οικείς για να καλύψουν τις σχέσεις των εμιράτων με τους τζιχαντιστές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τα um Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι ένα ομοσπονδιακό κράτος το οποίο αποτελείται από 7 Εμμυράτα τα οποία όμως είναι αυτόνομα. Ε, έχουν μεγάλα από θέματα πετρελαίου, αλλά εμεράτα αντλούν ε, τον πλούτο τους από ε, ναυτιλιακές ε, δραστηριότητες και πολύ συχνά επιδίδονται σε παράνομες χρηματοπιστωτικές ε, δραστηριότητες, απάτες με το ΦΠΑ, ξέπλυμα χρήματος κλπ πάσης φύσεως εγκληματικές δραστηριότητες τις οποίες ε, επιδίδονται τα κράτη αυτά. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα το οποίο να αφορά ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια και να δίνει τη δυνατότητα συνεργασίες με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για την πάταξη αυτών των εγκληματικών φαινομένων είναι απαραίτητο να υπάρξει μια θεσμική συνεργασία με τις χώρες της εγγύη και της Μέσης Ανατολής για να αποτελέσει τη βάση του κοινού αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Αλλά βεβαίως χρειαζόμαστε κάποιες ποιοτικές υψηλής ποιότητας δομές αυτής της συνεργασίας οι χώρες του κόλπου από τη μία συνεργάζονται με τη Δύση αλλά από την άλλη ε, τρέφουν στους κόλπους τους ε, φονταμενταλιστές και μελλοντικούς ε, τρομοκράτες. Και πολύ συχνά θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου που δεν θα είναι δυνατόν να συγκαλύπτεται αυτού του είδους η υποκριτική τακτική και να προωθεί τη συνεργασία με τέτοιου Τα Εμμυράτα είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτής της ε, πρακτικής και ελπίζω να χρησιμεύσουν σαν ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Η Επιτροπή Γιουρεβά, κυρία Πρόεδρο, η Επιτροπή σημειώνει το αίτημά του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου για να υποστηριχθεί η σύναψη συμφωνίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα αποτελέσει αυτή η συμφωνία το πρώτο βήμα για μια ανισχυμένη συνεργασία για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, ιδιαίτερα χρηματοοικονομικής φύσεως. Υπό τις παρούσους, παρούσες συνθήκες και με δεδομένη την ε, γεωπολιτική αστάθεια της περιοχής, η σύναψη της συμφωνίας αυτής ελπίζουμε να σημαίνει σημαντικά πλεονεκτήματα σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αντιμετώπιση της ε, σοβαρή εγκληματικότητα. Ωστόσο, στο σημείο 4 θα θέλαμε να σχολιάσουμε το ψήφισμα του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για την ε, κανονισμό της Europol. Συμφωνήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει τις συνθήκες που αφορούν ε, την ε, τα προσωπικά δεδομένα και την διαβίβαση προσωπικών δεδομένων με τρετές χώρες από τη Europol. Η συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν περιλαμβάνει την ε, διαβίβαση τέτοιων προσωπικών δεδομένων και έτσι ελπίζουμε να... Μάλλον πιστεύουμε ότι το σημείο 4 δεν ε, ταιριάζει στο ψήφισμα. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ε, λίγη συζήτηση.